Αν δεν διαφωνείτε, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 9 του κανονισμού, θα διαβιβάσω στον ενδιαφερόμενο την απόφαση αυτή. Στις 6 Φεβρουαρίου 2014 αποφάσισα τον κύριο Γκότφριντ Πλούμ, σύμφωνα με το άρθρο 153.3 μικρό α, να ε, τον επιπλήξω. Ε, αμέσως ε, ενημερώθηκε και στις 12 Φεβρουαρίου έλαβα την επιβεβαίωση της παραλαβής ε, αυτού του ε, θέματος. Και πάλι σύμφωνα με το άρθρο 153.1 ενημερώθηκαν και οι πρόεδροι της Επιτροπής ΕΚΟΝ και ΦΑΜ. Ε, έχει 15 μέρες ο κύριος Μπλουμ για να προβάλλει ένσταση. Την Τετάρτη, σύμφωνα με το άρθρο